Uh, Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Περιμένω να καθίσετε. Καλώς ορίζουμε με χαρά τον Επίτροπο Κατάινεν για τον ε, δομημένο διάλογο. Ευχαριστούμε που ήρθατε λοιπόν. Ξέρουμε ότι πάντα διατηρείται καλές επαφές με την Επιτροπή μας. Υπάρχουν θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Και θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο για να μην χάσουμε άλλο χρόνο για την, για την παρουσίασή σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. θα επικεντρωθώ στην ε, κυκλική οικονομία και τα συναφή ζητήματα. Καθώς αναμένονται προτάσεις στις αρχές του επόμενου έτους για την κυκλική οικονομία. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που συνιστά ορόσημο στο δρόμο για μια οικονομία με λιγότερες εκπομπές άνθρακα Άλλωστε πιστεύουμε ότι θα πρόκειται και για μία από τις κύριες εξελίξεις για το μέλλον, όπως η ψηφιοποίηση ή η ρομποτοποίηση. Και έχουμε ήδη υιοθετήσει τις βασικές γραμμές, τις κύριες πρωτοβουλίες τις υιοθετούμε στους επόμενους μήνες και αφορούν τα πλαστικά, την αποσύνδεση της παραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα, τον περιορισμό των πλαστικών και των αποβλήτων τους και άλλα. Και βέβαια ορίζουμε δείκτες για, τον υπολογισμό της πρόοδου της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη Τρίτον, θα έχουμε μία πρόταση νομοθετική για την ε, εξεργασία αστικών λιμάτων. Τέταρτον, πολιτικές επιλογές για τα χημικά και τα απόβλητα. Πέμπτον, τα απόβλητα ως στήριγμα της κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν κάνουμε διαβουλεύσεις για να συλλέξουμε τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων. Μια σειρά από, δια... από ε, δημόσιες διαβουλεύσεις έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει πλατφόρμες δημόσιες για να ευνοηθεί ο διάλογος όπως η παραδείγματι χρηματοδότηση των αποφυλητών τροφίμων ή της ε, ε απώλειας τροφίμων, της ε, σπατάλης τροφίμων καλύτερα, έχει ανοίξει ήδη. Και θα ήθελα ξεκινώντας να αναφερθώ στη στρατηγική για τα πλαστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ετοιμάσει την στρατηγική αυτή για το τέλος του έτους. Εξετάζει μια σειρά από μέτρα, νομοθετικά, οικονομικό μέτρο, μέτρα υποστήριξης, αλλά και δημοσιονομικέ δεσμεύσεις. Είναι τεράστια σημασία βέβαια η βιομηχανία του πλαστικού στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έχει πολλαπλές εφαρμογές σε σχέση με την κυκλικότητα. Μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για καινοτομία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η χρήση και η απόρριψη των πλαστικών αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται, δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. γιατί τα περισσότερα πλαστικά, ενώ θα είχαν τη δυνατότητα να μπουν στην κυκλική οικονομία, απορρίπτονται ή πηγαίνουν στους αποτεφρωτήρες ή καταλήγουν σε χωματερές ή στους ωκεανούς. Πράγμα το οποίο συνιστά σοβαρό πρόβλημα και για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία. Και γιατί στην οικονομία έχει αντίκτυπο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα το θέμα αυτό. Η στρατηγική λοιπόν θα προτείνει νέα καινοτομία και επενδύσεις ως τη λύση για την αντιμετώπιση του πλαστικού ως αποβλήτου για την ένταξη του στην κυκλική οικονομία και αυτό βέβαια μέσα στο πλαίσιο και της αναθεώρησης της Γενικής ε, Νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα και ταυτόχρονα με τη στρατηγική αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που θα συμπληρώνει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030. Οι διεθνείς πτυχές της διαχείρισης των πλαστικών αλλά και η επέκταση του σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι μεγάλο και σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας αυτού του μοντέλου. Θα κρυθεί δηλαδή το μοντέλο μας από την εφαρμογή, από την εισαγωγή του πρωτύπου της κυρικυκλής οικονομίας για τα πλαστικά και από άλλες χώρες, γιατί μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε έτσι και πρόσβαση σε ε, δευτερεύουσες αγορές πρώτων υλών. Ενθαρρύνουμε ή θα ενθαρρύνουμε την ε, επαναχρησιμοποίηση των ε, λιμάτων κατά τρόπον ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες σε νερό με δεδομένη τη σπάνιδα των υδάτινων πόρων και εδώ έχουμε προτάσεις για, τις, για τη γεωργική άρδευση ώστε να αξιοποιείται να αξιοποιούνται τα λύματα ε, όπου είναι δυνατόν και οικονομικό. Στην οδηγία για το πόσιμο νερό τώρα, έχουμε μια οδηγία για το πόσιμο νερό, προχωρούμε στην αξιολόγησή της, προσπαθούμε να εισαγάγουμε όρους οικονομικούς χρήσης του πόσιμου νερού, σημαντική απώλεια πόρων προέρχεται από διαρροές στα δίκτυα που φτάνουν και στο 23% του πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές ποιότητας με βάση και τα επιστημονικά στοιχεία της Παγκόσμιας Οργανώσης Υγείας θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο νερό της βρύσης και θα μειώσει την κατανάλωση νερού από μπουκάλια, πλαστικά και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας μέχρι το τέλος του έτους. Η χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας. Επιχειρηματικά μοντέλα όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας θα χρειαστούν νέους χρηματοδοτικούς πόρους και μέσα το Ευρωπαϊκό Ταμείο βέβαια για τις στρατηγικές επενδύσεις αλλά και το αντίστοιχο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι λύσεις αλλά θεωρούμε ότι θα χρειαστεί μια νέα πλατφόρμα που θα εστιάζεται συγκεκριμένα στην κυκλική οικονομία και γι' αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, τον Ιανουάριο του 2017 ιδρύσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή μια πρώτη πλατφόρμα για την κυκλική οικονομία που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μεταβούν προς την κυκλική οικονομία διευκολύνοντας την παραγωγή και τη χρηματοδότηση, τη γένεση και τη χρηματοδότηση προϊόντων κυκλικής οικονομίας. Έγινε μια δεύτερη ανακοίνωση τον Οκτώβριο είχαμε τη δεύτερη ανακοίνωση το Σεπτέμβριο του 2016 για την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης και την αναγέννηση του χρηματοδοτικού συστήματος ε, που είναι απαραίτητη για να υλοποιηθούν οι οικονομικοί μας στόχοι αλλά και οι περιβαλλοντικοί μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το πακέτο μέτρων της κυκλικής οικονομίας για το περιβάλλον. Και έτσι τώρα ε, προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε το χρηματοδοτικό σύστημα κατά τρόπο βιώσιμο. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πρώτη και εντυπωσιασμένοι μπορώ να από την πρώτη έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την ε, ε, λειτουργία του συστήματος της, της πλατφόρμας δηλαδή. Περιμένουμε και τα τελικά συμπεράσματα στο τέλος του έτους. Η βελτιωμένη νομοθεσία για τα απόβλητα όμως συνιστά τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση, διαχείριση των, ε, στη βελτίωση σε οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς όρους. Είναι όρος ε, απαραίτητος βεβαίως γι' αυτό. Υπάρχουν, δυνατότητες, υπάρχουν ανάγκες για σοβαρά κίνητρα που θα βοηθήσουν τη μετάβαση στην ε, κυκλική οικονομία. Έχουμε περάσει μέσα από διαπραγματεύσει αρκετά δύσκολε, αλλά βλέπουμε και πολλά ανοίγματα και δυνατότητε διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ένα πεδίο κοινό στο οποίο πρέπει να χτίσουμε και μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να διαδραματίσει το ρόλο του διαμεσολαβητή για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εχθές, κυρίες και κύριοι, κάνατε μια συζήτηση εις βάθος για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και ενώ δεν θα είχα να προσθέσω ιδιαίτερα στο όσο υπόθηκαν εχθές, επιτρέψτε μου μερικά λόγια για το πολύ επίκαιρο αυτό θέμα. Αυτή τη στιγμή μα απασχολούν τα προσεχή βήματα ύστερα από την αντίρρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικό με τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στο πλαίσιο τη νομοθεσία για τα ζυζανιοκτώνα. Μα αποστέλλει ένα σαφέ μήνυμα με την αντίρρησή του του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, λέγοντά μα ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν τα επιστημονικά κριτήρια όπω τα είχε ε, υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, θέλουμε να βρούμε μια λύση, γιατί έχουμε δει αρκετέ καθυστερήσει το να μην υπάρξει λύση θα ήταν κακή λύση για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλους μας. Δεν μπορούν να διατηρηθούν τα προσωρινά κριτήρια κατά τρόπο βιώσιμο είτε για τη δημοσία είτε για το περιβάλλον. Αυτό το δεχόμαστε όλοι και οι εμπλεκόμενοι φορεί. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηριχθεί σε μια ορθολογική, σε μια λογική προσέγγιση. Την είχαν υποστηρίξει τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι δεν έχουμε μεταξύ μα τόση απόσταση στο να βρούμε λύση. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μια εκδοχή που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή για το Συμβούλιο όπω και για το Κοινοβούλιο και επί τη ευκαιρία απευθύνω έκκληση για συνεργασία από πλευρά σας στην προσπάθεια αυτή. Αλλά επιτρέψτε μου αγαπητοί και κύριοι βουλευτές να σας υπενθυμίσω ότι κατά την έγκριση των κριτηρίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το πρώτο ρυθμιστικό σύστημα στον κόσμο που θα έχει νομικά δεσμευτικά κριτήρια που θα προσδιορίζουν τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τι σημαίνει, τι είναι ενδοκρινικός διαταράκτες και που θα, τον εντοπισμό, θα επιτρέπει τον εντοπισμό τους μέσα στο, ε, στα ζυζανιοκτώνα. Είναι τεράστια η ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Μετά τη συζήτηση μαζί, μας, θα, μαζί μου σήμερα θα συζητείτε τα κριτήρια ε, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες τα βιοκτώνα. Η Επιτροπή είναι στη διάθεση για να σας προσφέρει κάθε απαραίτητη διευκρίνηση με την ελπίδα πάντα ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μία διέξοδο, μία λύση ώστε οι ενδοκρινικές και οι διαταράκτες να βρουνε να καλυφθούν από την νομοθεσία. Κυρίε και κύριοι, σταματώ εδώ. Είμαι στη θέση σας και εάν είναι δυνατόν θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, για αυτή την συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων σας σε σχέση με την Επιτροπή μας. Όλα αυτά που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά για μας και προσβλέπουμε σε περαιτέρω προτάσεις και στρατηγικές για τα πλαστικά, για την χρηματοδότηση βιώσιμων προγραμμάτων κλπ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κωνσταντινός του ΕΛΚ πρώτα. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσατε. Δεν είμαστε και πολλοί που σας ακούσαμε, να ξέρετε όμως ότι εκτιμάμε την τακτική σας παρουσία στην Επιτροπή μας. Όταν μας παρουσιάζετε δηλαδή τις στρατηγικές της Κομισιόν, μιλήσατε ευρέω για τη στρατηγική αυτή και τις φιλοδοξίες της στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Χαίρομαι που προβλέπονται διάφορα μέτρα για την κυκλική οικονομία που παρουσιάσατε λεπτομερώς, μαζί με, βέβαια με τη στρατηγική για τα πλαστικά που με βρίσκει σύμφωνη και την οποία ελπίζω να λάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε επίσης και στους διαταράκτες, στους ενδοκρινικούς, αλλά υπάρχει κάτι που με λυπεί, δηλαδή ότι απουσιάζει πλήρως η υγεία από αυτή τη στρατηγική. Μεταξύ των διαφορών τομεακών μέτρων που αναφέρθηκαν, κανένα δεν αφορά ξεκάθαρα το, τη βιομηχανία της υγείας, γιατί είναι μια βιομηχανία με μεγάλη προστομινή αξία που έχει τροποποιήσει, έχει μεταμορφώσει η ψηφιακή οικονομία, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την οικονομία μας αλλά και για την υγεία των ασθενών. Για ποιο λόγο λοιπόν υπήρξε αυτή η παράληψη και πώς θα την προτίθεστε να δώσετε μια συνέχεια στο στρατηγικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας των φαρμακευτικών προϊόντων που αναφέρθηκε σε ανακοίνωση της Κομισιόν του 2012 με τον τίτλο «Μία πιο ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία υπέρ της ανάκαμψης και της ανάπτυξης». Καταλήγω λέγοντας ότι χαίρομαι που βλέπω πούμε ότι στη χώρα μου τώρα μάλιστα τη Δευτέρα είχαμε τέσσερα προγράμματα που έλαβαν το πράσινο φως από την Κομισιόν για 100 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Για αυτά λοιπόν τα προγράμματα που έγιναν δεκτά, πείτε μου, υπάρχει στόχευση προς συγκεκριμένα προγράμματα. Ποια είναι αυτή η στόχευση, να μας πείτε. Και να μου πείτε επίσης ποιο τμήμα αυτών των προγραμμάτων αφορά συγκεκριμένα την ενέργεια του περιβάλλον σε σχέση με το σύνολο των προγραμμάτων που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το σχέδιο Γιούνκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγε η πρόεδρο. Η κυρία Ντάλεκ, μέρο των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστώ τον κύριο Κατάινεν που ήρθε σήμερα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που σχετίζονται και που αναφερθήκατε, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Το πακέτο για τα πλαστικά πρώτα. Αν και κακή οικονομία το πακέτο αυτό και η στόχευση στα πλαστικά. Αναφερθήκατε σε κάποιες διεθνείς πτυχές που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές κι εγώ, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αναλάβει μόνη της η Ένωση, όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Παρ' όλα αυτά, τι σχέδια έχει η Κομισιόν ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις διεθνείς πτυχές και να πάει παραπέρα. Σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν κάποια έγγραφα που διέρευσαν σχέση με τη στρατηγική και φαίνεται ότι η Κομισιόν χρησιμοποίησε τον όρο TAF αυστηρός για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Επίσης, επίσης σε σχέση με αυτό, μιας και είστε υπεύθυνο και αρμόδιος για ανάπτυξη και σταθερότητα, στις αρχές του χρόνου εσείς είπατε στις Βρυξέλλες ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται στην πρωτοπορία της καινοτομίας και της ανανέωσης όσο αφορά την καθαρή ενέργεια σε σχέση βέβαια πάντοτε με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τις ε, δεσμεύσεις που έχουμε υπό την COP21. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση φαίνεται να μένει πίσω όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Βλέπετε να επενδύουν οι χώρες, μέλη, ώστε να βρίσκονται ακριβώς στην πρωτοπορία της καινοτομίας και της έρευνας και η πλατφόρμα αυτή που λέγαμε έχει συγκροτηθεί ώστε να καλύψει την έλλειψη χρηματοδότησης αλλά να προσελκύσει επίσης και πιο κοινοτόμες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, εσείς μιλήσατε για σχέδια, για φιλοδοξίες, για προθέσεις κλπ. Να σας πω ότι τα σχέδιά μας και οι προθέσεις μας θα πρέπει να προσαρμόζονται στις πραγματικές πιθανότητες υλοποίησης. Η κατάσταση νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά κάποια προϊόντα για τα οποία θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα μάλιστα στα πλαίσια μιας οδηγίας. Η Κομισιόν μάλλον η Επιτροπή μας είχε πιο φιλόδοξη ε, σχέση ή συγγνώμη στάση σε σχέση με αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα όπως ας πούμε αυτά που αφορούν το κάδμιο. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι η ψηφορία θα είναι και κάπως δύσκολη στην Ολομέλεια επειδή ε, στην Επιτροπή η ψηφοφορία ήταν ε, στο αποτέλεσμα πολύ κοντά. και υπάρχουν διάφοροι που έχουν άλλες θέσεις, δηλαδή θέλουν κάποιοι να υπάρχουν περιορισμοί στα όρια και μάλιστα κάποιες χώρες δεν έχουν δικιά τους παραγωγή ή έχουν περιορισμένη παραγωγή. Άλλες χώρες θέλουν να περιορίσουν την παραγωγή ανάλογα με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Όλη αυτή η σύγκρουση τέλο πάντων που αφορά αυτό το θέμα των λοιπασμάτων αφορά την υγεία. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία. Δεν υπάρχουν τεχνολογικές Οπότε ίσως στην ουσία να έχουμε να κάνουμε απλά και μόνο με σύγκρουση συμφερόντων. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω μήπως εσείς θεωρείτε ότι στο Συμβούλιο θα μπορούσε να σχηματιστεί, να δημορφωθεί μια οριστική θέση μέχρι τα τέλη του χρόνου. Είναι υπαρκτή αυτή η δυνατότητα. Και η Κομισιόν έχει πρόθεση να διευκολύνει τη λήψη αυτής της απόφασης στο Συμβούλιο. Αν λοιπόν μια απόφαση είσαστε υπέρ της μείωσης του ορίου του καθμίου. Μια και χώρες με ελεγχούν συγκεκριμένε απόψεις. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, βέβαια υπέρ κάποιων συγκεκριμένων χωρών μελών, οι οποίες θα αποκτήσουν κάποιο πλεονέκτημα ενδεχομένω. Μήπως ήταν καλύτερο αντίθετα να έχουμε μία θέση η οποία θα διευκολύνει την ίσως στην αγορά και άλλων λοιπασμάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κοίταζα την οθόνη να δω κατά πόσο ξεπεράσατε το χρόνο. Γκέρ Μπράντι, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κατάινεν, για αυτή την επισκόπηση για το τι μπορούμε να αναμένουμε από την Κομισιόν του επόμενου μήνε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, η στρατηγική για τα πλαστικά. Προσβλέπουμε στην πρόταση βέβαια της Κομισιόν και ρωτάω στοχευμένα αν ενημερώνομαι σωστά φαίνεται ότι υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στην Κομισιόν για τα μικροπλαστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Βλέπουμε να υπάρχουν όλο και περισσότερε αποδείξει ότι αυτά τα μικροπλαστικά είναι παντού. Υπάρχουν πολλέ χώρε με οι οποίε έχουν εκφράσει ανησυχία. Οπότε το ερώτημά μου προ εσά είναι το εξή. Έχετε πρόθεση να δώσετε μάχη για την ε, θέσπιση πολύ αυστηρών πολιτικών σε σχέση με τα μικροπλαστικά. Ας πούμε η χρήση των μικροπλαστικών στα καλλιντικά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω εσείς τώρα πρέπει να αποφασίσετε αν θα το περιλάβετε αυτό ή όχι. Δεύτερη ερώτηση, ένα ζήτημα που δεν αναφέρατε αλλά που είναι στο χαρτοφυλακείο σας, η βιοποικιλότητα. Πριν χρόνια είχαμε την κατάσταση της φύσης από την από το περιβαλλοντική υπηρεσία και όλα τα στοιχεία είναι ενισχυτικά ότι δηλαδή δεν κάνουμε ό,τι πρέπει για να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2020 στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής και η Κομισιόν βεβαίως ε, σοφά αποφάσισε να μην ανοίξει την οδηγία για τα πτηνά και ε, τα ενδιατήματα αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε βεβαίως τους στόχους της βιοποικιλότητας αλλά όχι μόνος τους, όχι χωριστά. Είδα πάρα πολλά στοιχεία από την έρευνα, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας, ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά για να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί. Αλλά μας είπε ο συνάδελφός σας, ο Επίτροπος, να περιμένουμε τις επόμενες ε, προοπτικές, γιατί η τωρινή πολιτική για τη γεωργία θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι επιπτώσεις στη φύση. Οπότε ρωτάω ξεκάθαρα, εσάς. Μπορούμε να αναμένουμε σύντομα σχετικά μία δήλωση από την Κομισιόν να πει δηλαδή ότι συγγνώμη, κάνουμε ό,τι μπορούσαμε, δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ή αντίθετα, μπορούμε να αναμένουμε μία νέα όθηση από την Κομισιόν, μία νέα στόχευση, μία νέα εστίαση ώστε να πετύχουμε ακριβώς αυτούς τους στόχους βιοπικιλότητας του 2020. Αλλιώς θα κάνουμε το ίδιο όπως την προηγούμενη φορά, θα καταλήξουμε στο ότι δεν θα τους πετύχουμε και θα πούμε εντάξει, θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά και μετά θα περνάνε τα χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Λοιπόν, τι μπορούμε να προσδοκάμε από σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια, ο Σέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, η κλιματική αλλαγή που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και ο αντίκτυπο θα οδηγήσει σε ε, κοινωνικές και οικονομικέ απώλειες τι οποίε δεν μπορούμε να φανταστούμε καν σήμερα ε, και θα υπάρξουν και αναρρύθμιτα ανθρώπινα θύματα. Η μόλυνση για παράδειγμα του υδροφόρου ορίζοντα με ζυζανιοκτώνα και ε, τοξικέ τοξικές χημικές ουσίες όπως και η αύξηση των σκουπιδιών γενικότητα και των απορριμμάτων, η αύξηση των εκπομπών διοξιδίου, καταστροφή ε, των τροπικών δασών. Είναι όλα προβλήματα. Ε, και ε, φέτος έχουμε για δεύτερη φορά την τον εορτασμό τη ε, ημέρα σε ό,τι αφορά τι αλλακτικές Ε, Ο πληθυσμό ε, τη Βιλού ε, αυξάνεται τόσο γρήγορα και δαπανά σε τόσο μεγάλο βαθμό του υφιστάμενους πόρου, σαν να μην υπάρχει μέλλον. Και τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε αυτή την τελευταία, στα τελευταία 100 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτή η αιμονή με την οικονομική ανάπτυξη τελικά δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσε λύσει προσφέρει για την ευημερία των ανθρώπων και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποιον ο οποίος ε, πιστεύει ότι με την αηφόρο οικονομική ανάπτυξη, με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη ε, θα έχουμε πραγματικά ένα βιώσιμο μέλλον. Δηλαδή, να πιστεύει κανείς κάποιο τέτοιο, ε, κάτι τέτοιο είναι αφελής ή είναι τρελός. αυτή η κατάσταση τελικά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια, ε, οδηγήσει περισσότερε σε σειράξει. σειράξεις. Και ε, βέβαια η, ε, το να επαφέμαστε στα, στα πλαστικά δεν αποτελεί μια λύση για αυτό το πρόβλημα της κατασπατάληση των πόρων. Δεν θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το σημείο εκείνο όπου θα έχουν κατασπαταληθεί όλοι οι φυστάμενοι πόροι μας. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μα. Ε, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της φυστάμενης γενιάς, της σημερινής γενιάς, χωρίς ωστόσο να υπονομεύουμε το μέλλον των μελλοντικών γενιών. Ε, και ένα και μόνο ερώτημα θέλω να σας ε, θέσω. Ποια είναι η δική σας άποψη ή τι θα νομίζατε αν θα ήταν σωστό δηλαδή ε, να αλλάξουμε το οικονομικό μας ε, μοντέλο ανάπτυξης έτσι ώστε να έχουμε την ε, σωστή και δίκαιη κατανομή των πόρων η οποία θα διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στον, στον κόσμο μας σήμερα και θα ήθελα και σας ευχαριστώ των προτέρων για μια δίκαιη και τίμια και ειλικρινή απάντηση. ο κύριος Κρέκ. Ευχαριστώ. Ε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, για την περιουσία σας σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το σύστημα τη κυκλητής οικονομία. Ε, Κάνοντα αυτή λοιπόν τη μετάβαση προς την κυκλητή οικονομία, αντιλαμβανόμαστε όλο ένα και περισσότερο καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και αποτελεί βέβαια ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το ζήτημα λόγω των, των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν στα διαφορετικά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση των σχετικών για την ανάκτηση των σχετικών πρωτονινών. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, παρότι υπάρχει και μια... Δεν υπάρχει τόση μεγάλη βούληση από την ε, πλευρά ε, των κρατών μελών. Ε, και μόνο ένα μικρό ποσοστό τη χρηματοδότηση γίνεται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Άρα λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξή θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπου χρήση αυτών των δευτερευουσών πρώτων υλών όταν θα έχουμε εφαρμόσει στην πράξη αυτά τα ανακυκλωμένα υλικά. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε καύση πολύτιμων τέτοιων πρώτων υλών, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τι απαραίτητε δυνατότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επαναχρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ενισχυμένε επενδύσει σε αυτό το τομέα. Περισσότερα λοιπόν κονδύλια θα πρέπει να δαπανιστούν σε αυτή την αναχρησιμοποίησή του. Και δεν θέλουμε να εξάγονται αυτά, αυτές οι πρώτες ύλες σε τρίτες χώρες, γιατί βέβαια συχνά η περαιτέρω επεξεργασία του γίνεται, γίνεται με ακατάλληλους τρόπους και με περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικά δυσμενείς ε, επιπτώσεις. Οπότε τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση. Ε, και ένα τρίτο ερώτημα αφορά την ε, σταδιακή για τα πλαστικά της Ένωσης. Αναμένουμε δηλαδή μια σταδιακή σταδιακή από την Επιτροπή στα τέλη αυτού του έτους. Ε, εδώ έχετε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη και την τρίτη ε, γενιά των ε, πίστοξ για τα πλαστικά. Λέτε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για τον τομέα της ενέργειας και αλλού. Μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν περαιτέρω προτάσεις δράσεων των της Επιτροπής προκειμένου να είναι δυνατή η καλύτερη χρησιμοποίησή τους για να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, ολοκληρώθηκε τώρα ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων, οπότε πρωτού ακούσουμε τα περαιτέρω ερωτήματα των συναδέλφων, να δώσουμε το λόγο στον πρώτο κατάλληλο για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω απαντώντας τα ερωτήματα της κυρία Κροστέτ. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τη υγεία, Η Επιτροπή εξάγει μία σειρά από δράσει στον τομέα τη υγεία προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε αυτό το τομέα. Ε, και πολλέ από αυτέ τι στρατηγικέ αποτελούν βέβαια συνέχεια υφιστάμενων ε, διεδράσεων. δράσεων. Υπάρχουν ε, ωστόσο και τρει νέε πρωτοβουλίε. Καταρχήν, έχουμε την ψηφιοποίηση της υγειονομικής ε, και πρόνοιας Συγκεκριμένα προετοιμάζουμε μια ανακοίνωση η οποία προβλέπει συγκεκριμένα βήματα για την υποστήριξη των κρατών μελών για αξιοποίηση περισσότερων ψηφιακών μέσων ε, σε, στον τομέα της υγείας, δημιουργία δηλαδή περαιτέρω, ε, υποδομών, υποστήριξη ε, των πολιτών και ούτω καθεξής. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτή η πρωτοβουλία θα έχει αντίκτυπο τόσο στον κλάδο της υγείας, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέψει για πιο ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, θα μειώσει ε, και το, τις δαπάνες ε, λειτουργίας, επιχειρησιακές δηλαδή δαπάνες ε, των τομέων Επίσης, θα προβούμε σε μια αξιολόγηση της νέων τεχνολογιών. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε εδώ ε, τα νέα καινοτόμα ε, φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και ε, ιατρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στον τομέα. Και στην επιστολή Προθεσίστου, ο πρόεδρο Γιούνκερ αναφέρθηκε σε ένα σχέδιο δράση ό,τι αφορά του εμβολιασμού. Ε, θέλουμε δηλαδή να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη ε, να αυξήσουν του ε, στατικέ εμβολιασμού προκειμένου να προληφθούν κρούσματα ασθενειών και με αυτόν τον τρόπο βέβαια ισχυθεί και η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν ω προ το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Τώρα, από εκεί και μετά αναφερθήκατε στι επενδύσει που σχετίζονται με το περιβάλλον. Εδώ τώρα θα αναφερθώ στα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ. Ήδη το ΕΦΣΥ έχει χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό αριθμό επενδύσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Επίσης κάποια μεγάλα project κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα στον τομέα του χάρτου και του χαρτοπολτού, έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΥ. Δηλαδή σε αυτές τις επενδύσεις οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει τον τρόπο εμ, λειτουργίας τους, όχι μόνο προς την παραγωγή του χαρτιού, αλλά εφαρμόζοντας και περισσότερα στοιχεία κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή αξιοποιούν περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη φάση της παραγωγής, αλλά και τα υποπροϊόντα παραγωγής ε, χάρτου, αξιοποιούνται ε, ως προϊόντα που μπορούν να μεταπολίθουν. Άρα λοιπόν αυτές οι επενδύσεις έχουν γίνει μέσω του ΕΦΣΙ. Τώρα, όταν θα εφαρμοστεί το νέο ΕΦΣΙ, το ΕΦΣΙ 2.0, θα έχουμε και ε, συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά επενδύσεις COP21. Ε, και προβλέπεται ότι το 40% αυτών των ενισχύσεων από το ΕΣΥ θα αφορούν τέτοια project από τη Συμφωνία ΔΕΚΟΠ21. Άρα λοιπόν το ΕΦΣΙ δείχνει πράγματι να είναι το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για ε, τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και ήδη έχει λειτουργήσει πολύ καλά, έχει επιφέρει καλά αποτελέσματα σε project σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και κάποια από αυτά έλαβαν χώρα στη Γαλλία. Τώρα, κύριε Αντάλη, αναφερθήκατε στις, ε, στη στρατηγική για τα πλαστικά και το πώς αυτή συνδέεται με τη γενική μας ε, στρατηγική. Ε, ο κύριος Τζέπαρντι αναφέρθηκε στο ζήτημα των μικροπλαστικών, οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω στα δύο αυτά ερωτήματα από κοινού. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλά ορισμένη στρατηγική για τα πλαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε και αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή αν βρούμε τρόπους να μειώσουμε την γενικότερη κατανάλωση πλαστικών, εάν μπορέσουμε να προβλέψουμε κάποιες, ε, ένα κανονιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα ε, πλαστικά από βιοαπόρριτα και αν μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε μία αγορά για δευτερεύοντα πλαστικά, secondary plastics, όλες αυτές οι νέες δράσεις, όλα αυτά τα πλαίσια θα εφαρμόσουν και για όσες επιχειρήσεις της αεροδαπής δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν θα υπάρξει αντίκτυπος και προς τα έξω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενθαρρυνθούν δηλαδή οι επιχειρήσεις και όλοι οι φορείς ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες και τον ίδιο τρόπο λειτουργίας που έχουμε μέσα. Ε, και αυτό θα το κάνουν δηλαδή και άλλες χώρες, οι αρμόδιοι φορείς τους. Και από εκεί και μετά θέλουμε να ε, εξαγάγουμε εντό εισαγωγικών αυτό το μοντέλο σε άλλε χώρε. Ειδικότερα σε χώρε εταίρου, σε στενή βέβαια συνεργασία μαζί του. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα διαδώσουμε τι πρακτικέ από την δική μα πλευρά. Ακριβώ για αυτό το λόγο ένα σωστό να χαράξουμε μια σωστή στρατηγική. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα των μικροπλαστικών, ναι, ασφαλώς θα αποτελέσει μέρος της ε, του σχεδίου δράσης μας. Ε, τα ψάρια δηλαδή γνωρίζουμε ότι είναι ήδη ε, γεμάτα από μικροπλαστικά, αλλά και τα ζήματα μας στα εδάφη μας είναι γεμάτα από ε, μικροπλαστικά, οπότε σίγουρα τα μικροπλαστικά θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου δράσης. Ε, κυρία Ντάλη, επίσης ε, έθεσε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και το κατά πόσο δηλαδή έχουμε προχωρήσει αρκετά εδώ και ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Ε, αληθεύει πράγματι αυτό που είπατε, ότι τα κράτη-μέλη δεν επενδύουν στο βαθμό που ελπίζαμε και στο βαθμό που είχε συμφωνηθεί προκειμένου να προωθηθούν εδώ οι κοινοτομίε. ωστοσο Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δίνουν έμφαση στην κοινοτομία και επίση το Horizon 2020 δίνει ευκαιρίε για τέτοιου είδου επενδύσει στην καινοτομία και μπορεί κανεί να δει τι μελλοντικέ στρατηγικέ για την κοινοτομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση από δύο πτυχέ. Καταρχήν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ε, ε, συστάσεις ανά κράτος μέλος σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή θα πρέπει να, δοθεί, να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση της ερεύνας, αλλά και περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης δηλαδή, για παράδειγμα κατάρτιση εκπαιδευτών. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να αναλάβουν τα στα κράτη-μέλη. Και μια δεύτερη διάσταση, μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι εάν πράγματι χρειαστεί να αναθεωρήσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τότε θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς εκείνους όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Και ελπίζω πως η καινοτομία και η έρευνα μαζί με τα ζητήματα ε, ασφαλείας είναι εκείνα όπου έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ προσωπικά λοιπόν θα πρότεινα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Ε, η κυρία Βυσνιεύσκα έθεσε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα και κατά πόσο τα επίπεδα καδμίου είναι αντιδειγμένα ή όχι. Θεωρώ πως θα πρέπει να παραμείνουν τα επίπεδα όσοι έχουν σήμερα, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση σήμερα για τα κρατημέλη. Εάν μειωθούν ε, τα επίπεδα ακαδημίου, είναι προφανώς θετικό για την ανθρώπινη υγεία και ε, ταυτόχρονα μπορούμε να προτρέψουμε την αγορά να προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε ό,τι αφορά τα σχετικά προϊόντα. Ε, με αυτόν τον ε, τρόπο νομίζω πως αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική η οποία θα βασίζεται στην παραγωγή λοιπασμάτων από τότε ε, με αυτόν τον τρόπο θα, ε, με αυτή την εφαρμογή, με, τα χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα καμία που θα προβλέπουμε, θα έχουμε θετικό αντίκτυπο. Ε, για παράδειγμα, τη μείωση του φωσφόρου, της χρήσης φωσφόρου στα λοιπάσματα. Λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη όλα τα γεωπολιτικά ζητήματα, παρόλα αυτά θεωρώ πως λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη το ε, ε, το τι επιτυγχάνουμε μέσω των μειωμένων ε, επιπέδων καδμίου, θεωρώ πως πράγματι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη στρατηγική και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη και να υπάρξει συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα, ο κ. Σάκη σε ένα σχετικό ερώτημα. Έχουμε ένα ε, σχέδιο δράση που περιλαμβάνει 15 ξεχωριστέ πράξει. Οι περισσότερε από αυτέ ελοποιούνται φέτος, οπότε πριν ε, από το τέλος ε, της ε, θητείας της Επιτροπής θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ως προς τα αποτελέσματά τους και από εκεί και μετά οι δράσει αυτέ προσανατολίζονται και προ ε, την ε, εκπλήρωση των στόχων που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά την απώλεια τη βιοπικιλότητα έω το 2020. Άρα λοιπόν, έως τα μέσα του 2020 θα έχουμε, κάνει και μια, έχουμε ετοιμάσει μια αξιολόγηση στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα και ο στόχος εδώ ο στόχος βέβαια θα είναι να ορίσουμε και τη μελλοντική στρατηγική για την προστασία της βιοπικιλότητας ε, από το 2020 και μετά. Αλλά και ε, το δίκτυο Natura των προστατευόμενων δηλαδή ε, περιοχών θα συνεχίσει να αποτελεί μια σταθερή βάση για αυτές τις μελλοντικές στρατηγικές προστασίας της βιοπικιλότητας. Ο κύριος Σεκ έθεσε ένα θεμελιώδες ερώτημα ως προς το κατά πόσο έχει νόημα το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης και ως προς το εάν θα έπρεπε να αναπτύξουμε ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο. Πρόκειται προφανώ ε, για ένα πολύ ιδεολογικά φορτισμένο και θεμελιώδες ερώτημα. Αλλά κατά τη δική μου άποψη δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα μπορούσε μια μηδενική ή πολύ ε, ασθενή ανάπτυξη να μα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στόχων μα ε, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Για παράδειγμα, Ε, αν δούμε κάποια μοντέλα τα οποία αντίστοιχα δηλαδή έχουν εφαρμοστεί για παράδειγμα στην ε, Βενεζουέλα, στην Κούβα ή στη Βόρεια Κορέα θα δούμε ότι δεν είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει δηλαδή η ανάπτυξή μα να είναι ανταγωνιστική και γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, υποστήριξη απέναντι στην ε, αηφόρο ακριβώ ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και νομίζω πως ε, όταν αναφερόμαστε σε αυτόν τον όρο κυκλική οικονομία και το επίθετο κυκλική και ουσιαστικό οικονομία έχουν νόημα. Δηλαδή προφανώς και το οικονομικό στέλος είναι σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει σε, αυτήν την, σε αυτόν τον κυκλικό χαρακτήρα που έχει αυτή η οικονομία να δημιουργούνται και κέρδη. Τέλος, τέθηκε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τη σχετική χρηματοδότηση. δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Καταρχήν, έχουμε το ζήτημα της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Εάν καταφέρουμε να θεσπίσουμε νομοθεσία που θα θέτει δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη, θα δημιουργούσαμε σημαντικά κίνητρα για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και πιο αεφόρων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Δηλαδή μια τέτοια νομοθεσία θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στα κράτη-μέλη και στις περιοχές τους ως προς το πώς να διαχειριστούν καλύτερα τις ε, ροές ε, των αποβλήτων που διαχειρίζονται. Ε, το πρόβλημα σε αυτό το τομέα δεν είναι κυρίως οικονομικό. Γιατί ε, όταν έχουμε, εφαρμόζουμε τέτοιε ε, στρατηγικέ, ε, αναγκάζονται οι σχετικοί τομέ να προσαρμοστούν, να, να υιοθετήσουν δηλαδή εναλλακτικά μοντέλα. Αλλά ήδη 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται στα διαρθρωτικά μας ταμεία για τη βελτίωση ακριβώ των συστήματων διαχείριση αποβλήτων στα κράτη-μέλη. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή είναι μία και μόνη οικονομική ρόλη. Και για το 2018 έως 2020 έχουμε προβλέψει 860 εκατομμύρια ευρώ για τις καλύτερες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. Δηλαδή η σχετική τεχνολογία ήδη υφίσταται σήμερα. Υπάρχουν για παράδειγμα εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που αξιοποιούν για παράδειγμα κοπριά ε, ζώων. Και εδώ ακριβώς έχουμε ένα σύστημα το οποίο και δημιουργεί προσθεμένη αξία από αυτή την κοπριά και ταυτόχρονα προστατεύει τα εντροβό μας όλες τα ύδατά μας. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και το μέλλον για την βιομηχανία λιμασμάτων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων τώρα. Ένα λεπτό η κάθε ερώτηση τώρα πια. Η κυρία Σούρτσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κατάιναν για να εξασφαλιστεί η κυκλική οικονομία και οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων. Ε, θεωρούμε ότι θα υιοθετηθούν τα απαραίτητα νομοθετήματα και ότι δεν θα είναι αυτό το τέλος της ιστορίας, αλλά η αρχή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια απαριθμεί συγκεκριμένα αδικήματα κατά του περιβάλλοντος και σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την δυνατότητα ενίσχυσης του ρυθμιστικού και διοκτικού συστήματος. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό διαφθοράς ορισμένα κράτη-μέλη και μπορεί αυτό να επηρεάσει την ε, τήρηση των ανωτέρων στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διατυπώσει τα αντίστοιχα μέτρα ή εργαλεία για την τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου και νομοθετικού πλαισίου. Δεύτερη ερώτηση. Με πιο θετική προσέγγιση έχουμε το εκατομμύρια νέε θέσει εργασία, η ενίσχυση της, ε, του θεματολογίου για τι δεξιότητε των νέων αλλά και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη είναι λύσει που απευθύνονται στου νέου. Θα έχουν μακροπρόθεσμη όμως, ε, μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασία στα διάφορα κράτη-μέλη και έσκοπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία παρουσιάσουν πολύ ψηλά ποσοστά ανεργία, πολύ ψηλότερα από ό,τι στα άλλα, τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανεργία. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, θα κάνει κάτι η Επιτροπή, κάποιο εργαλείο θα ετοιμάσει για να ισοσταθμίσει την κατάσταση. Κυρία Βαλάν, δύο ρωτήσεις δηλαδή είχατε. Μάλιστα, είχα δύο ρωτήσεις για σήμερα. Λάινεν. Πολύ σωστά είπατε κύριε κύριε Αντιπρόεδρε, ότι η κυκλική οικονομία είναι ένα τιτάνιο έργο. Έχει να κάνει με την μεταμόρφωση της οικονομίας μας. Οδηγεί στη μεταμόρφωση της, ε, τη μεταμόρφωση της οικονομίας μας. Βεβαίως είναι ε, και σημείο των καιρών πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους σπόρους μας. Ξέρω ότι είχατε πάει και στην Κίνα, είχατε επικοινωνία και επαφές με την ε, μεγάλη αυτή χώρα. Είχα πρόσφατα εδώ σε μία ε, διάσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία ήρθαν και οι Κινέζοι ε, μου είπανε λοιπόν ότι και στο θέμα της κυκλικής οικονομίας σε 5-6 χρόνια θα μας έχουν ξεπεράσει γιατί κάνουν σοβαρές επενδύσεις. Οικοσχεδιασμός λοιπόν, οικολογικός σχεδιασμός. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Έχει πολλά να αποκομίσει κανείς από τη διαμόρφωση ενός προϊόντος. Αν είναι καλή η διαμόρφωση του προϊόντος, ο σχεδιασμός του σωστός, ε, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του, μπορούμε ακόμα και να αποφύγουμε τελείως τα απόβλητα. Οικολογικός σχεδιασμός λοιπόν, τι κάνει η Ευρώπη γι' αυτό. Μεγάλο δυναμικό κρύβεται πίσω από αυτόν και πιστεύω ότι και η βιομηχανία στην Ευρώπη είναι έτοιμη να ε, αναλάβει τα σχετικά βήματα. Thank you very much. Uh, Κυρία Βυσνιεύσκα. Monsieur Pagnier. Euh, monsieur le Commissaire. Ο κύριος Παγνιού, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι ξεκινώ κύριε Επίτροπε με ένα μεγάλο Μπράβο για την προσέγγιση ευρύτατη και πολύ ε, σαφή του θέματος των ενδοκρινικών διαταρακτών που ακούσαμε στην αρχή της τοποθέτησής σας ε, και το Κοινοβούλιο γενικότερα αλλά και εμείς ειδικότερα ως Επιτροπή Περιβάλλοντος βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η προσπάθεια και οι αγώνες μας ε, στέφονται με επιτυχία γιατί να εσείς εδώ αντιπρόεδρος και στο υψηλότερο επίπεδο της ε, ιεραρχίας για τα θέματα της ε, υγείας, της δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχίστε και μας μιλάτε για ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μπράβο σας και συγχαρητήρια. Ωστόσο, για την... Ε, σπατάλη τροφίμων, ένα θέμα για το οποίο δεν τοποθετηθήκατε καθόλου. 89 εκατομμύρια τόνοι σπαταλώνται από τρόφιμα. Είναι τα τρόφιμα που πετάμε κάθε χρόνο στην Ευρώπη και μπορεί αυτό να φτάσει και στους 120 εκατομμύρια τόνους το χρόνο για την Ευρώπη μόνο. Είναι ανεύθυνη αυτή η απουσία σχεδιασμού και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν στόχο περιορισμού της πατάλης των τροφίμων για 30% έως το 2025 και 20% για το 2030, όπως υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2017. Αυτή την πρόταση λοιπόν θέλω να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποστηρίζει. Φλόρεντς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε την Και σήμερα και χθες άκουσα με προσοχή τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις. Μπορώ να υπογραμμίσω με ιδιαίτερη έμφαση τα όσα υπόθηκαν για την οδηγία πλαίσιο. Η χώρα μου έχει παραπευθεί στο δικαστήριο και σωστά νομίζω. Ακούω βέβαια από τους ε, συναδέλφους εδώ ε, ότι μου λένε πράγματα τετριμένα και για το θέμα της προστασίας των υδάτων. Βεβαίως έχουμε θέμα προστασίας των υδάτων, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την παρουσία φαρμάκων στα ύδατα. Τι κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό το οποίο ίσα ίσα ψελίζουν ορισμένοι. Η Πολωνή συνάδελφος που δυστυχώς απεχώρησε τίκα. Αλλάξτε παρακαλώ τη στρατηγική σας. Ε, μην αλλάξετε τη στρατηγική σας για το θέμα της ε, ε, χρήσης λιπασμάτων. Είπε ο κύριος Γερμπράντε ότι είναι επιστημονικό επίτευγμα η χρήση λιπασμάτων στην ε, ε γεωργία. Το να αυξηθούν τα επίπεδα του καδμίου αποτελεί ε, οπισθοδρόμηση Εν πάση περιπτώσει, α σταματήσουμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δώσουμε εξηγήσει στου καταναλωτέ μα γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Ντόν. Εδώ, πρόεδρε, στα αριστερά. Για του ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης έχουμε ακούσει πολύ ωραία λόγια και γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Ε, ε, πολύ ωραία λόγια λοιπόν από την Επιτροπή, πλατφόρμα ε, με συμμετοχή πολλαπλών εμπλεκομένων φορέων για τον Ιανουάριο, ανακοινώνεται πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά για τι θέσει εργασία, τι συγκεκριμένα έχει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει πρόοδο στον πολιτικό, τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό ε, τομέα, αλλά και στη διακυβέρνηση και επίση η χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού στην επόμενη 7 ετία, πώ θα στοχευθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασία και τι ρόλο μπορεί να δραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία συνεργασία και διαλόγου με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, γιατί ξέρουμε ότι θα εμπλακούν οι κοινωνικοί φορείς, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ε, από πλευράς της Επιτροπής. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κυρία Ντουλάη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα επιμένω στην ερώτηση του συναδέλφου Παγνιού για τη σπατάλη τροφίμων. Πρόταση μεθοδολογική για τον υπολογισμό της σπατάλης τροφίμων. Πότε θα έχουμε. Γιατί δεν αρκεί να ζητούμε μείωση ποσοστιαία, αλλά χρειάζεται και ένας ορισμός μεθοδολογία για να αξιολογηθεί τι είναι αυτή, η, τι συνιστά σπατάλη. Κυρία Σέρπιρκ. Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση που αφορά την, ε, τις κατοχώρες. Βιοαέρια, πράσινη, ενέργεια. Πώς πάνε και τα πράγματα, καλά, μας πείτε κάτι. Είστε εξοικειωμένο με την υπόθεση, γιατί ξέρω ότι έχουν μείνει πολλές εκκρεμότητες. Η Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Ο Επίτροπος. Περιβαλλοντικά αδικήματα καταρχάς. Οι ένωμες μας τάξεις αντιμετωπίζουν ε, διαφόρων τύπων αδικήματα. Η Επιτροπή δεν έχει μεριμνήσει, δεν έχει υπόψη τη δημιουργία ειδικού αδικήματος, διόνομα αδικήματος σχετικού με το περιβάλλον. Η κατηγορία αδικημάτων. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας, όντως υπάρχει πολλή διαφθορά. Αλλά δεν, κάνουμε δια... δεν διαφοροποιούμε μεταξύ των διαφορών κατηγοριών αδικημάτων, ώστε να προτείνουμε την εισαγωγή ιδιαίτερων μέτρων για κάθε συγκεκριμένο τύπο. Η δίωξη των εγκλημάτων είναι πάντα στα χέρια των αρχών, κατά κύριο λόγο στα χέρια των αρχών των κρατών μελών. Υπάρχουν συζητήσεις για την ανάληψη μεθόδων βέλτιστων πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, όπου υπάρχουν εγκλήματα ε, κατά του περιβάλλοντος. Απασχόληση. Απασχόληση είπατε ότι διαφέρει πολύ μεταξύ κρατών μελών. Οι τάσεις είναι πάντως προς την αντιστροφή αυτής της ε, ισορροπίας. Έχουμε την υψηλότερη απασχόληση. Η ανεργία έχει πέσει στα επίπεδα του 2008-2009 Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν συνθήκες και κατάσταση χειρότερη από ό,τι κάποια άλλα ή ότι δεν υπάρχουν ομάδες ευάλωτες ή νέοι επί παραδείγματι ή άλλες που ε, δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό ε, κοιτάει τέτοιες αιτήσεις ε, μελέτες ανάπτυξης, τέτοιες ε, συστάσεις κατά κράτος, τη διαδικασία του εξαμήνου, αλλά και άλλα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας, μέσα που έχουμε στη θέση μας για να συμβάλλει στην αντιστροφή του φαινομένου. Σας διαβεβαιώ ότι έχουμε πληθώρα ευκαιριών να στήριξουμε τα κράτη-μέλη, αλλά μεταρρυθμίσεις στη θέση των κρατών μελών δεν μπορούμε να κάνουμε όταν αυτές χρειάζονται. Πάντως σταθεροποιείται η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσωτερική αγορά είναι πρόσφορη στην δημιουργία ένδοσης συνεργασίας, ε, παραγωγικότητας ανταγωνισμού και εμπορίου. Ο κύριος Λάριν μίλησε για την Κίνα. Κίνα μπορεί να σταθεί εταίρος καλός για μας στην κυκλική οικονομία, γιατί έχει, έχουν ανάγκη να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουν τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκονται περισσότερο από ότι εμείς, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Αλλά επειδή ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση, ή να το πω αλλιώς, η Κίνα μπορεί να είναι μια μεγάλη αγορά για τις ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να αναπτύξουμε μια κοινή αγορά, ε, μια μεικτή μάλλον αγορά για την, ε, μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοια προϊόντα και λύσεις. Η κυρία ενδιαφέρεται για την κυκλική οικονομία και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από του τομεί του οποίου θα μπορούσε δυνάμει να αναπτυχθεί η συνεργασία μα. Είχαμε αποκλίνουσε απόψει σε διάφορα σημεία με την Κίνα, αλλά η κυκλική οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντο είναι θέματα στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Ο οικολογικό σχεδιασμό, και ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Εμεί ακολουθούμε πρακτικές λύσεις στο θέμα αυτό. Κοιτούμε ε, προϊόντα που θα είναι και διαλειτουργικά και πιο βιώσιμα με λιγότερα απόβλητα και κάνουμε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς για το τι θεωρούν σκόπιμο. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να καλύψει περισσότερες διαστάσεις της οδηγίας του οικολογικού σχεδιασμού. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό πολύ. Η διαλειτουργικότητα, παράδειγμα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους Ευρωπαίους. Η δυνατότητα παραδείγματι να αντικαταστήσει κανείς το τζάμι του τηλεφώνου του αν του σπάσει. Αυτό είναι αδύνατο σχεδόν. Ε, όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συγκεκριμένες βέβαια υποσχέσεις αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας δώσω για τις αλλαγές που θα έχουμε υποβάλει μέχρι το τέλος της θητείας μας, αλλά θα κάνουμε προτάσεις. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι εξαιρετικό εργαλείο και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη ενίσχυση της αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας και όπως πολύ σωστά επισημάνατε γίνεται δεκτό από την βιομηχανία. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα ότι ίσω είναι το πιο παρεξηγημένο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ότι αλλάζει σιγά σιγά η διάθεση απέναντι στην οδηγία, γιατί έχει αρχίσει ο κλάδος να συζητεί τα θέματα αυτά μαζί με τους οργανισμούς των πολιτών, των καταναλωτών, πολύ πιο ανοιχτά τα θέματα του οικολογικού σχεδιασμού. Ε, σπατάλη τροφίμων, με δύο ερωτήσεις. Και εδώ πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο έχουμε απευθυνθεί στους εμπλεκόμενους φορείς, έχουμε στήσει τις απόψεις τους γιατί θέλουμε να αντιληφθούμε σε ποιο επίπεδο ε, είναι σκόπιμο να υπολογίζεται η σπατάλη των τροφίμων. Από πού προέρχεται δηλαδή αυτή η σπατάλη τροφίμων. Από τη γεωργία, από την την ε, βιομηχανία, το λιανικό, το χονδρικό εμπόριο, τα εστιατόρια, από ποιους τομείς και πώς θα μετράτε η σπατάλη τροφίμων και η ροές αποβλήτων τροφίμων. Όταν αντιληφθούμε τις διαστάσεις του φαινομένου, τότε μπορούμε να προτείνουμε λύσεις. Αλλά πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ε, πόσες, είναι οι σπατάλοι τροφίμων και από πού προέρχεται. Για τον κύριο Φλόρεντς. τα φάρμακα στα ύδατα. Μα ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να εισαγάγουμε κανονισμό που να καλύπτει τα θέματα της παρουσίας του καδμίου. Και βέβαια για τα λοιπάσματα έχουμε αντίστοιχες προθέσεις. Η πρωτοβουλία για τα την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε προδιαγραφές ή να γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι πράγματι ασφαλές ε, το νερό αυτό για, την, ε, για τον άνθρωπο. Για την ε, οδηγία, για τα λοιπάσματα. Αυτά που έχουν χαμηλότερο επίπεδο καδμίου, γιατί υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι αυτά τα οποία μπορούν να πολλούνται ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Όποιος θέλει μέσα στην επικράτειά του να χρησιμοποιεί άλλου, άλλης περιεκτικότητας λοιπάσματα, μπορεί μόνο μέσα στην επικράτειά του. Αλλά εμείς θέλουμε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερως για το υγρά λοιπάσματα ή ε, για αντίστοιχες λύσεις. Έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά. Ίσως καλό θα ήταν κάποια στιγμή να εξηγώ και στο Συμβούλιο τι ακριβώς διακυβεύεται εδώ, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, ότι είναι τόσο δύσκολο να λυθεί. Αναφερθήκατε στην βιώσιμη ανάπτυξη, τους στόχους, ε, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να κοιτάξω όχι μόνο και να το μετρήσω από τη σκοπιά των βιώσιμων, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και σε κάθε τι, είτε πρόκειται για κυκλική οικονομία, είτε πρόκειται για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται με τον ίδιο γνώμονα. Γιατί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα από κάθε μορφή πολιτικής. Και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται σε όλες τις πλατφόρμες, τις σχετικές με, το, με τους στόχους ε, που φέρουν τον τίτλο «Πλατφόρμα για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης», αυτό δεν θα σημαίνει ότι έχει αποκλειστεί το Κοινοβούλιο, γιατί στην πραγματικότητα συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τις προτάσεις για το βιοαέριο είναι κομμάτι της ε, πρότασης για, την, ε, για τα βιοκαύσιμα. Ε, θα είναι και στο μέλλον. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε τεχνολογία, την καινοτομία και τι περαιτέρω βέβαια εξελίξεις της τεχνολογίας. Αλλά υπάρχει και η άλλη διάσταση και το άλλο ζήτημα, το πόσο καλά έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες σε τοπικό επίπεδο. Άρα θέλει και ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις. Πάντως το βιοαέριο θα έχει σημαντικό ρόλο στις πράσινη, στην πράσινη οικονομία και στη διαχείριση των αποβλήτων στο μέλλον. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Πολύ θα ήθελα να συνεχίσετε αυτή τη συνεργασία και οποτεδήποτε έχετε κάτι να συζητήσετε μαζί μου, είμαι στη θέσή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, President, for... Ευχαριστώ πολύ, Αντιπρόεδρε, που ήρθατε σήμερα. Βασιζόμαστε σε εσά για να συνεχίσουμε και την ισχυρή σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Έχουμε και ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών μέχρι να ξεκινήσουμε τις πληροφορίες. Hello, everyone. Let's start with the votes. Ας ξεκινήσουμε με τις ψηφορίες. Ποια είναι η πρώτη? We start with the vote on... Uh, Ξεκινάμε. Κυρία Κροστέτ, αξιολόγηση αναλογικότητας πριν από την έγκριση νέας ρυθμίσης των επαγγελμάτων. Παρακαλώ, οι παρατηρητές να κάνουν στοιχεία και να παρατηρούν μόνο. Πρώτα λοιπόν έκθεση της κυρίας Γκροστέτ. Αξιολόγηση τη αναλογικότητας πριν από την έγκριση νέας ρύθμισης των επαγγελμάτων. Θα ψηφίσουμε μαζί μια ομάδα, μια δέσμη τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ διακόπτη πρόεδρος 62 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 τώρα 66 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά θα ελέξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Και πάλι. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71. 73 73 Πάμε στο 73, στο σημείο. 73 υπέρ. Κατά, άποχες, απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά, άποχες, απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω, αλλά να ελέξουμε, γιατί δεν μου ήταν ξεκάθαρο. 87. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται μαζί οι 92 και 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά 98 ξαναλέει ο πρόεδρος υπέρ 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 106 πάμε λέει πρόεδρος. 5. Όχι 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 106 και 107 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται.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 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει πρόεδρος να ελέγξουμε, ωραία ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας γελάει η πρόεδρος τυχερή μου να λέει αλλά έκρινα από την στάση της ομάδας, αλλά φαίνεται ότι ήταν μικρή η πλειοψηφία. 116 ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ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 Κατά. Α, ένα όπλο λέει πρώτος. Ο, ο είπε. Υπέρ. Υπέρ τη 16. Ποιος είναι υπέρ τη 16. Κατά. Αποχέ. Να το ελέξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Περάς. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Καταπίπτει. 24. Υπέρ. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ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 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48, 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέξουμε. 48. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Και τώρα πέρας. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά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 Τελική ψήφος ηλεκτρονικά. Άρχεται. Και τώρα πέρα. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην συγκήτρια. Επόμενο σημείο. Η έκθεση της κυρίας Τσάλτερς ε, εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στατιστικής για τα άτομα με αναπηρία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 49 άρχεται ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 48 υπέρ κατά ψηφίσαμε ήδη για τη 48 Οπότε 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή μάλλον να ελέγξουμε την τροπολογία 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 56. Πέραση της ψηφοφορίας και απορρίπτεται η 56. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 τμηματική πληροφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε τροπολογία 6. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα επί του συνόλου της έκθεσης ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται και τα συγχαρητήριά μας στην εισηγήτρια. Επιτάνει τη ε, γενοτομίε του τομέα τη καθαρή ενέργεια. Εισηγητή ο κύριο Σεκ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται.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 Εγκρίθηκε. Η 11. Όχι. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. So I see right and left split it completely on this one. That's, uh, <laughs> that was the secret. Mm, χωρίστηκε η αριστερά από την δεξιά από ό,τι φαίνεται. Μάλλον η δεξιά μεταξύ της και η αριστερά μεταξύ της. Εγώ παρακολουθώ τα χέρια των συντονιστών, αλλά ψηφίσατε διαφορετικά. 12 κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ. Απόχειας απερίφθη. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά Το ΕΛΚ δεν το βλέπω να κινείται. 23 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Η 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχεται πέρας και εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει And it is closed. Πέρας. Και εγκρίνεται συγχαρητήρια. Επόμενο. Επισκόπηση περιβαλλοντικής, υλοποίηση περιβαλλοντικής πολιτικής ε, με τους συνεισηγητές και αρχώ, αρχίζω με την 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 28 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 σε δύο τμήματα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απερίφθης δεύτερο υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε. Και η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 46 υπέρ κατά αποχές απερίφ... εγκρίνεται λέει πρόεδρος 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 69 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ. Δεν ψηφίζουμε, όχι. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 75 υπέρ κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. Να και δυσκόνετε το χέρι σας. 75 και πέρας. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. 76 αλφα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη μόνο ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ. Απερίφθη η πρώτη. Μπέλεψα τα λόγια μου. δύο υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 6 δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 7 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 8 και 15 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε τη 16 and it's closed it is adopted Seven... και εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ Close. Πέρας. Και εγκρίνεται συγχωρητήρια. Next uh, and last uh, action plan for nature. Τέλος, το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία. Με πέντε συνεισηγητές επίσης. Τροπολογία 8 πρώτα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, λέει η πρόεδρος. Να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά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 εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε λέει πρόεδρος. Για το πρώτο τμήμα της 39. πέρας και εγκρίνεται λέει πρόεδρος. 39 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. 73. Καταπίπτει έτσι. Καταπίπτει. 73. Οπότε δεν την ψηφίζουμε. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 να ελέγξουμε την 55 ας το ξανακάνουμε ας ξαναψηφίσουμε 55 ποιος είναι υπέρ Α, καλά, εντάξει, ας πάμε τότε στην ηλεκτρονική ψήφο. Ελέγχουμε για την 55. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 καταπίπτει. 75 τότε. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές 81 υπέρ και να το ξανακάνουμε πάλι πρώτος 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήταν το πέμπτο τμήμα λέει η πρόεδρος τώρα έκτο τμήμα της 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές θα ξαναψηφίσουμε λέει πρόεδρος 87 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104-105 ομού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τεσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Άρχεται. Και τέλειωσε η ψήφος. Τέρμα, λέει η Πρόεδρος. Εγκρίνεται, τελειώσαμε τις πληροφορίες και τελειώσαμε και τη μέρα μας κιόλας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά πότε. Την ερχόμενη εβδομάδα 19 του Οκτώβρη λέει η Παρακαλώ τους συντενιστές να μείνουν για να κάνουμε τη συνεδρίασή μας.